τη συνεδρίαση είναι διαθέσιμα. Υπάρχουν παρατηρήσεις για τα πρακτικά. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις για τα πρακτικά. Και έτσι θεωρείται ότι κυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης. Κάποιες παρατηρήσεις για την έναξη της συνεδρίασης. Σήμερα είναι η μέρα της Ευρώπης. Πέρασα το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σήμερα στην Φλωρεντία